διώξουν έτσι ώστε να έχουμε πραγματικά ε, βιώσιμα σχέδια τα οποία να αποφύγουν την ε, κερδοσκοπία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την εισηγήτρια. Κλείνοντας τη συζήτηση, θα ήθελα να πω ότι είμαι πολύ υπερήφανος για την πρωτοβουλία σου και ο παππούς σου πέρασε πολλά χρόνια στη φυλακή για να δώσει μεγάλη αγώνα, μεγάλο αγώνα κατά του φασισμού και χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι άξια συνεχιστής. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο στις 11.30. Το επόμενο θέμα είναι η δήλωση της Επιτροπής για τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή του Δούναβη και νομίζω ότι έχει προσέλθει, είναι εδώ ο Επίτροπος Σέπκοβιτς, ο οποίος και θα μιλήσει εξ ονόματος της Επιτροπής. Έχετε το λόγο. Χωρίς μικρόφωνο, ο Επίτροπος. Now it Ξεκίνησα με τη δήλωση ότι η στρατηγική του Δούναβ είναι πολύ σημαντική για την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί η περιοχή αυτή περιλαμβάνει 14 χώρες, 8 ε, κράτη-μέλη και 6 μη κράτη-μέλη με πολλά εκατομμύρια κατοίκους. Από τότε που εισήχθη η στρατηγική έχουμε πιστεί έτσι περαιτέρω για την αλληλεξάρτηση των κρατών αυτών και για το πόσο μπορούν να υποφεληθούν από την ε, βελτιωμένη συνεργασία συνεργασία και το συντονισμό των εργασιών τους. Διαπιστώσαμε πώς είναι δυνατόν να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητά τους αν ε, γίνουν από κοινού πράξη στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, της αγοράς εργασίας, της παιδείας και της ασφάλειας. Και γνωρίζουμε επίσης πολύ καλά ότι η περιφέρεια του Δούναβη είναι το αντικείμενο ε, των δύο τελευταίων γύρων της διεύρυνσης και τώρα προσπαθούμε με τη στρατηγική αυτή να προσεγγίσουμε και τους νέους ε, υποψηφίους από τα Βαλκάνια. Όπως γνωρίζετε αυτή η στρατηγική παρουσιάστηκε από την Επιτροπή τον Απρίλιο του 2011 και στηρίζεται σε τέσσερις πυλώνες. Τη σύνδεση της περιοχής του Δούναβη, προστασία του περιβάλλοντος, οικοδομώντας στην ευημερία και ενίσχυση της περιφέρειας του Δούναβη, το πώς έχουμε προχωρήσει, που φτάσαμε σε αυτό τον ένα χρόνο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή συντάσσει την πρώτη έκθεσή τους η οποία θα υιοθετηθεί στις αρχές του 2013. Θέλω όμως να σας κάνω μια πρώτη παρουσίαση της ε, πρώτης αυτής αξιολόγησης. Όπως ξέρετε, ο συνάδελφός μου, ο Επίτροπος Χάν, ταξίδεψε στην περιοχή αυτή και συμμετείχε σε διάφορες ε, δράσεις που ξεκίνησαν χάρη στη στρατηγική του Δούναβη. Είναι σαφές ε, ότι χάρη σε αυτή τη στρατηγική εμφανίστηκε μια νέα δυναμική, νέα συνεργασία σε διάφορα επίπεδα. Οι πολιτικοί παράγοντες, το επίπεδο των επιχειρήσεων ή η κοινότητα της ε, έρευνας. Για πρώτη φορά διαπιστώσαμε ότι οι χώρες προσπαθούν να βρουν κοινέ λύσεις στις κοινέ δυσκολίες τους. Η στρατηγική αυτή ταχύτατα γίνεται μια πλατφόρμα για μια μακροπρόθεσμη συνεργασία. Αυτό που θα είναι πολύ σημαντικό για το μέλλον είναι το πώς θα συντονίσουμε τις εθνικές πολιτικές με την ευρωπαϊκή στρατηγική. Σαφώς αυτό πρέπει να, ε, πρέπει γίνει ε, μετά, με τον τρόπο που είπαν οι Υπουργοί ε, Μεταφορών οι οποίοι δεσμεύτηκαν με συγκεκριμένο τρόπο για τη βελτίωση της κατάστασης του Δούναβη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βοηθάει προσφέροντας νέες δυνατότητες για την ανανέωση του στόλου του Δούναβη να γίνει πιο σύγχρονος και πιο πράσινος με, τρόπο, με τρόπους βοή, παροχής βοήθειας προς τους ερευνητές. Γίνεται μια, ε, δημιουργείται ένα πρόγραμμα βελτίωσης των, της λήψης αποφάσεων και της συγκέντρωσης ε, περιβαλλοντικών στοιχείων στο Δούναβι. Η αστυνομική συνεργασία γίνεται βασική προτεραιότητα των κρατών μελών της περιοχής του Δούναβι. Και βεβαίως δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι μπορούμε να προωθήσουμε το τον τουρισμό με το όνομα του Δούναβη. Αυτά είναι λίγα από τα παραδείγματα. χθε. ο Επίτροπος Χάν ε, εγγενίασε την νέα γέφυρα μεταξύ ε, στη Ρουμανία και πρέπει να πω ότι αυτό είναι το δεύτερο άνοιγμα, το δεύτερο πέρασμα σε ένα σύνορο 600 χιλιόμετρων θα υπάρξουν πολλά διακρατικά έργα γιατί έχουμε πάνω από 50 έργα τα οποία είναι υπό εξέταση αυτή τη στιγμή ως έργα της, περιοχής του, της περιφέρειας του Δούναβη και τώρα περιμένουν για υποστήριξη και χρηματοδότηση. Το θέμα της χρηματοδότησης είναι φυσικά κρίσιμο, βασικό για την περαιτέρω επιτυχία. Η στρατηγική διαπερνά τις διάφορες πολιτικές της Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Προσπαθούμε λοιπόν να εισάγουμε το στοιχείο της μακροπεριφέρειας στο πλαίσιο της μελλοντική μας μακροπρόθεσμης στρατηγικής προγράμματα εταιρική σχέση που θέλουμε να δούμε πώ μπορούν να εφαρμοστούν και στα πλαίσια αυτά τη περιφέρεια του Δούναβη. Θέλω να υπενθυμίσω ότι έχει ξεκάθαρα ζητήσει το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αξιολογηθεί η έννοια της μακροπεριφερειακής στρατηγικής μέσα στο 2013. Αυτό θα είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για να δούμε πόσο επιτυχημένη είναι αυτή η αντίληψη. Εν κατακλείδη θέλω να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πολύ σημαντική δουλειά του και την υποστήριξη στα τεχνικά ζητήματα της στρατηγικής του Δούναβη. Το εκτιμούν πολύ και οι, αυτοί που την έλαβαν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Αντιπρόεδρο Σεύκοβιτς. Το λόγο έχει στο γύρο των πολιτικών ομάδων ο κύριος Ματούλα εξ ονόματος του ΕΛΚ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, η εξέλιξη της κρίσης μας δείχνει ότι υπάρχει αλληλένδετος χαρακτήρας των αγορών και γι' αυτό δεν μπορούμε παρά να λάβουμε υπόψη ότι ο κατακαιρματικός δεν βοηθάει. Χρειάζεται ενωμένη Ευρώπη, περισσότερη Ευρώπη. Ο πρόεδρος Μπαρόζο την προηγούμενη εβδομάδα στο Βουκουρέστι είπε ότι έχουν, έχει γίνει πρόοδος αλλά όχι επαρκής. Θα πρέπει να προωθήσουμε την πολιτική better spending η στρατηγική υπέρ του Δούναβη θα βοηθήσει στην σύγκληση και την ανταγωνιστικότητα. Οι προκλήσεις είναι πολύ μεγάλες και γι' αυτό χρειάζονται μέτρα εξέχοντος χαρακτήρα για να προωθήσουμε συγκεκριμένες πολιτικές υπέρ των παραποτάμιων περιοχών σε πολλά επίπεδα. Θα πρέπει να υποβοηθήσουμε και την μεταφορά εμπορευμάτων και προς τρίτες χώρες. Έτσι θα προωθήσουμε και την ανταγωνιστικότητα των παραδουνάβιων περιοχών, μειώνοντας τις οδικές μεταφορές και δημιουργώντας απασχόληση. Βεβαίως υπάρχουν και θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς τα οποία θα έπρεπε να προωθήσουμε στις παράκτιες περιοχές του Δούναβη. Θα πρέπει να προωθήσουμε και αυτές τις επιμέρους στρατηγικές. Χτες ο Επίτροπος Χαν είπε ότι χρειάζεται μία μεγαλύτερη συνδεσιμότητα διότι ε, πρόκειται για μια πολύ μεγάλη έκταση και για να είναι η στρατηγική επιτυχής θα πρέπει να άρουμε τα προσκόμματα τα οποία δεν επιτρέπουν αυτή τη συνδεσιμότητα. Τέλος, θα ήθελα να σας υποβάλω ένα, ένα ερώτημα. Ε, αν δεν υπάρχουν επιπρόσθετα χρηματοδοτικά μέσα, δεν θα μπορέσουμε να προωθήσουμε αυτή τη στρατηγική. Θεωρείται ότι θα πρέπει να αναθεωρηθεί η πολιτική της Επιτροπής επί του θέματος αυτού, έτσι ώστε να δοθεί μια νέα δυναμική. Θεωρεί ότι η Επιτροπή, η Επιτροπή ότι θα πρέπει να υπάρξει άμεση προσβασιμότητα, ιδιαίτερα ως προς τον διασυνοριακό χαρακτήρα του εγχείρηματος. Ο κύριος Σταμπάτζη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Νομίζω πως ε, είναι θετικό το ότι ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής, ο κύριος Σεύκοβιτς, έκανε δήλωση ενώπιον του Κοινοβουλίου για την στρατηγική του Δούναπη. Η Ουγγρική Προεδρία προφανώς ασχολήθηκε με το θέμα και ένα από τα μεγαλύτερα επιτευγματά της ήταν κάτι το οποίο καλωσόρισαν όλες οι ενδιαφερόμενες χώρες. Αυτό το οποίο χρειάζεται λοιπόν είναι συνεργασία. Είναι θετικό το ότι έχουμε επιτέλους μια στρατηγική του Δούναβη που επιτρέπει στενότερη συνεργασία μεταξύ των χωρών που βρέχονται από το Δούναβη ε, όσον αφορά τις μεταφορές, ε, ναυτιλία, τουρισμό κτλ. Αλλά πρέπει πρώτα απ' όλα να είναι πλεύσιμος ο ποταμός και οι χώρες βεβαίως οι οποίες διατρέχει πρέπει να καταβάλουν κάθε προσπάθεια και η Ουγγαρία αλλά και η Σλοβακία, ε, <clears throat> Ρουμανία ε, όλες πρέπει να χρησιμοποιήσουν και το νερό του με τρόπο κατάλληλο. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα πάρα πολύ μεγάλο δυναμικό το οποίο δεν έχει χρησιμοποιηθεί και νομίζω πως είναι πάρα πολύ καλό το ότι έχουμε μεταρρύθμιση της κοινής γεωρικής πολιτικής στο δεύτερο πυλώνα και χαιρόμαστε για το ότι θα έχουμε νέα κονδύλια διαθέσιμα για το σκοπό αυτό. Είναι πάρα πολύ θετικό αυτό για όλες τις χώρες ε, τις οποίες δεν τρέχει ο Δουναβής. Θα ήθελα να πω ότι ο κύριος ε, Ταμπάτζη έλαβε το λόγο εξ ονόματος των σοσιαλιστών, εξ ονόματος των φιλελευθέρων και για δύο λεπτά το λόγο έχει ο κύριος Τόιρερ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Το Κοινοβούλιο στήριξε με τρόπο ενεργό τη στρατηγική αυτή. Έχουμε το δίκτυο του Δούναβη με 60 βουλευτές, ε, γι' αυτό χαίρομαι για το ότι βρίσκεται το θέμα αυτό σήμερα στην ημερήσια διάταξη. Οι εξελίξεις όπως η γέφυρα μεταξύ Βιντι και Καλαφάτη είναι πάρα πολύ θετικές. Εγώ είχα την ευκαιρία να τις δω το καλοκαίρι, αλλά πηγαίνουν με ρυθμό σαλιγκαριού. Υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες. Ε, Δήμαρχοι στη Βουλγαρία λένε πως για να γίνει ένα έργο στο Δούναδη πρέπει να εμπλακούν 7 υπουργεία και άλλες χώρες ε, τις οποίες διατρέχει ο ποταμός έχουν την εντύπωση πως ε, στις πρωτεύουσε τους ε, παίζει δεύτερο ρόλο ο Δουναβής. Γι' αυτό ζητάμε από την Κομισιόν να γίνουν πιο συγκεκριμένα τα πράγματα και τα μέτρα. Στην τορνή προγραμματική περίοδο πρέπει να δοθούν μέσα για τη στρατηγική αυτή κονδύλια και στην επόμενη χρειάζεται μια ξεχωριστή γραμμή του προϋπολογισμού. Εδώ πέρα θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει και καλύτερη διοικητική ικανότητα να υποστηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να συνεργαστούν κέντρα μεταφοράς τεχνολογίας, αλλά πρώτα απ' όλα χρειάζονται και περισσότερες επαφές των πολιτών και διαπιστώνουμε πως πρέπει να υποστηριχθούν, αλλιώς δεν γίνονται. Εγώ έγραψα μια επιστολή στην καγκελάριο Μέρκελ και στον Επίτροπο τον κύριο Λεβαντόφσκι όπου πρότεινα μια επαφή των νέων του Δούναβη και με μια οικονομική στήριξη. Πάρα πολλοί νέοι ευχαρίστω θα έκανα αυτές τις, ε, τις επαφές αλλά δεν έχουν να πληρώσουν τα εισιτήρια κτλ. Ναι, και τα κοινοβούλια επίσης πρέπει να παίξουν έναν πιο ενεργό ρόλο και ελπίζω εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβουμε ηγετικό ρόλο και τα άλλα εθνικά και περιφερειακά κοινοβούλια να προσκληθούν για να προωθήσουμε ακόμη πιο ενεργά αυτή τη στρατηγική. Σας ευχαριστώ. Για τους ε, πράσινους, για δύο λεπτά, η κυρία Λόχμπίλερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Σεύκοβιτς, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι πάρα πολύ θετικό το ότι σήμερα έχουμε μια δήλωση από την Κομισιόν για την κατάσταση εφαρμογής της στρατηγικής του Δούναδη. Για εμάς τους βουλευτές δεν είναι πάντα ε, εύκολο να έχουμε πληροφορίες ε, οι οποίες είναι πρόσφατες. Και βεβαίως σημαντικό είναι και η εμπλοκή της κοινωνίας των πολιτών το οποίο πρέπει να γίνει ακόμα σε ορισμένες χώρες για την συνδιαμόρφωση της στρατηγικής του Δούναβη. Πώς θα γίνεται όμως αυτό εάν δεν είναι ενημερωμένοι εγκαίρως για τα πράγματα. Γι' αυτό σας παρακαλώ εσάς στην Κομισιόν μαζί με τις χώρες να καταβάλλετε περισσότερες προσπάθειες έτσι ώστε να ε, υπάρχουν εγκαίρως ή πληροφορίες για την εφαρμογή της στρατηγικής αυτής. Επίσης θα πρέπει να απαντήσετε περισσότερο, ε, να πρέπει να απαντήσετε σε μια γραπτή ερώτηση που έκανα με άλλους συναδέλφους ε, τον Ιούλιο του 2011 αφορά το θέμα της ναυσιπλοείας στον Δουναβή και συγκεκριμένα το κομμάτι που περνά από τη Βαβαρία μεταξύ Στράουφεν και Φίλσχόφεν ε, το οποίο, του οποίου η Κίτη θα αλλάξει και είναι ένα εξαιρετικό κομμάτι φύσης με διάφορα δάση τα οποία απειλούνται με καταστροφή από την αλλαγή της κήτης του ποταμού για να γίνει πιο πλέσιμο. Ο Επιτροπος Χάν είχε απαντήσει, αλλά όχι σε όλα τα μέρη της ερώτησής μας. Συγκεκριμένα δεν απάντησε στο ερώτημα, το οποίο ήταν ποια μέτρα θα λάβει η Κομισιόν για να διασφαλίσει διαφάνεια στα σημεία να λήψη αποφάσεων για να εγγυηθεί την ανεξαρτησία των εμπειρογνωμόνων. Ξέρετε πώ οι άνθρωποι εκεί πέρα αγωνίζονται για την ελεύθερη νευσυπλοεία του Δούναβη, γι' αυτό θα πρέπει να είναι σαφές το ποιοι μπορούν να επηρεάζουν την ανεξαρτησία των εμπειρογνωμόνων. Σας ευχαριστώ. Εξ ονόματος της Google, το λόγο έχει για ένα λεπτό ο συνάδελφος Αγκουράκης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε οι δράσει για την μακροπεριφέρεια του δούναβη δεν αφορούν την κάλυψη λαϊκών αναγκών όπω απασχόληση με δικαιώματα εκπαίδευση κατοικία πολιτισμό αντιπλημμυρικά έργα και έργα αξιοποίηση του υδάτινου πλούτου. η μακροπεριφέρεια δεν αφορά μια βιομηχανική και αγροτική ανάπτυξη με αυτά τα κριτήρια αλλά την εμβάθυνση τη ενιαία καπιταλιστική αγορά και των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων που έχουν οδηγήσει του λαού στην ανεργία τη μαζική φτώχεια και τη χρεοκοπία οι δράσει τη εξυπηρετούν την αντιλαϊκή στρατηγική Ευρώπη 2020 και του ενεργειακού κολοσσού ενώ αφαιρούν σημαντικού πόρου προ όφελο του σχεδίου διασυνδέοντα την Ευρώπη. Ο αναπροσανατολισμός και αξιοποίηση κονδυλίων τη πολιτική συνοχή θα ωφελήσει πρωτιστώ την κερδοφορία των επιχειρήσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που δρούν στι παγκόσμιε αγορέ, θα εντείνει το τσάκισμα των εργασιακών και λαϊκών δικαιωμάτων, θα οξύνει την ανισόμετρη ανάπτυξη γι' αυτό θεωρούμε ότι οι μεγάλοι χαμένοι θα είναι οι εργαζόμενοι που καλούνται με σκληρέ θυσίε να στηρίξουν μια ανάπτυξη που δεν αφορά τι ανάγκε του. Ευχαριστούμε. Τέλος, το λόγο ο κύριου Στάτλερ, ο οποίος θα μας θα μας μιλήσει ε, εξ ονόματος των μη εγγεγραμμένων. Ε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να επενδυμίσω πως η στρατηγική αυτή βασίζεται σε μια αυστρο-ρουμανική πρωτοβουλία. Η Αυστρία αντιλαμβάνεστε πως έχει μια ιδιαίτερη ιστορική εμπειρία. Δεν θα μπω τώρα στις λεπτομέρειες, θα ήθελα μόνο από το έγγραφο της ανακοίνωσης να αναφερθώ σε ορισμένα σημεία την προβληματική δηλαδή υποδομή, σιδηροδρομική, αεροπορική και λοιπά. Κοίταξα λοιπόν το τι προτείνεται όσον αφορά την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βλέπω μόνο Ευρώπη 2020. Ακριβώς αυτός ο τομέας που έχει ιδιαίτερη σημασία για τον χώρο αυτό θα αποτελούσε ένα πάρα πολύ προνομιούχο πεδίο δράσης για το πρόγραμμα συνδέοντας ε, την Ευρώπη και νομίζω πως ε, ακριβώς η αξιολόγηση αυτού του προγράμματος ε, θα μπορούσε να επικεντρωθεί στις ε, σιδηροδρομικές και λοιπές συνδέσεις γιατί εδώ πέρα υπάρχουν και τα απαραίτητα μέσα τα οποία μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και να κερδίσουμε πάρα πολλά για ολόκληρη την περιφέρεια και άρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έληξε ο γύρος εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων και θα περάσουμε στους επόμενους ομιλητές. Μαρία Γκαμπριέλ, τη συνάδελφο την οποία γνωρίζαμε ως κυρία Ναντελτσέβα και θα θέλαμε να την συγχαρούμε γιατί παντρεύτηκε και γι' αυτό ακριβώς άλλαξε και το όνομά της. Έχετε το λόγο κυρία Γκαμπριέλ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, χτες ολοκληρώθηκε η γέφυρα του Καλαφάτ. Όλοι οι επίσημοι αναφέρθηκαν στην στρατηγική του Δούναβη, η οποία θα βοηθήσει για να στην καλυτέρευση της ζωής των Ευρωπαίων. Πρέπει να δούμε τι έχει γίνει μέχρι τώρα, να σκεφτούμε τις προκλήσεις και το μέλλον. Πρέπει καταρχήν να σας υπενθυμίσω ότι εκατομμύρια Ευρωπαίοι περιμένουν τα αποτελέσματα αυτής της στρατηγικής. Το ίδιο και στη Βουλγαρία. Κάθε μήνα συναντιόμαστε με τους εκπροσώπους και το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης για να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους αυτής της στρατηγικής. Βλέπουμε την προσδοκά ο κόσμος. Δρόμους, λιμάνια, καθαρό νερό, τουρισμό, κέντρα νεότητας, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τι άλλο χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε την πολιτική θέληση για να εκπληρωθούν οι στόχοι αυτής της στρατηγικής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα σας στηρίξει κύριε Επίτροπε ξεκάθαροι όροι, ξεκάθαρες ε, ευθύνες. Και τρίτον, τρίτη ευθύνη είναι να είναι απλές οι διαδικασίες. Θέλω να επιστήσω την προσοχή σας στη συμμετοχή των νέων στη στρατηγική αυτή. Αυτή είναι η πιο δημιουργική, οι πιο καινοτόμη. Μπορούν να βοηθήσουν τη στρατηγική αυτή να πετύχει τους στόχους της. Δεύτερον, χρειαζόμαστε στρατηγική σε επενδύσεις. Υπάρχει το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Σε τι μπορούμε να στηριχτούμε κύριε Επίτροπε. Μόνο αν υπάρξουν επαρκείς πόροι, συντονισμένες δράσεις ε, και επενδύσεις στοχευμένες μπορεί αυτή η στρατηγική των τριών όχι να γίνει στρατηγική των τριών ναι. Ναι στις νέες ιδέες, ναι στις νέες επενδύσεις, ναι στην καλύτερη ζωή αυτών που ζουν στις ακτές του Δούναβη. Η κυρία Ντανσίλα έχει το λόγο για ένα λεπτό. Η συνεργασία στις παραδουνάβιες περιοχές ενισχύθηκε τα τελευταία χρόνια και Πιστεύω ότι η προσχώρησή μας ε, πρόωθησε αυτή τη ε, διαδικασία. Η στρατηγική του Δούναβη αποτελεί επαρκές ε, πλαίσιο για ανταλλαγές πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών στη λεκάνη του Δούναβη έτσι ώστε να ενισχύσουμε αυτή τη στρατηγική μόνο με ανταλλαγές πληροφοριών και ε, έρευνες σε σχέση με τη μόλυνση του Δούναβη θα, μπορούσαμε, θα μπορέσουμε να έχουμε μία σωστή διασυνοριακή διαχείριση έτσι ώστε να μην έχουμε μίζονες καταστροφές και μόλυνση του ποταμού. Θα πρέπει να προβούμε σε επαρκή χρηματοδότηση αυτού του βασικού σχεδίου. Ευχαριστώ. Gracias, Ευχαριστούμε. Για 1,5 λεπτό το λόγο έχει η κυρία Γιάνγκλη. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η στρατηγική του Δουναβή είναι ένα σημαντικό έργο με το οποίο αντιδράει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτά τα οποία θέλει ο λαός και ακριβώς ε, αυτή η θέληση του λαού εκδηλώνεται πάρα πολύ ε, ένεργα όσον αφορά και τη σύλληψη της στρατηγικής αυτής και μια προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω. Θεωρώ πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ πέρα ήταν κινητή ε, δύναμη και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να συνεχίσουμε να στηρίζουμε αυτά τα οποία θέλουν οι άνθρωποι. Δεν επιτρέπεται να εξαφανιστεί σε κάποιο σιρτάρι αυτή η στρατηγική. Πρέπει να μεταφραστεί σε συγκεκριμένα έργα. Γι' αυτό και η σημερινή σας δήλωση κύριε Επίτροπε έχει τόσο μεγάλη σημασία. Ο στόχος στρατηγικής είναι η ευημερία και η απασχόληση κατά μήκο του Δούναβη καθώς υπάρχει όσο και μεγαλύτερη δικτύωση και θα πρέπει να βρεθούν περισσότερο οι υποδομές και οι ανταλλαγές κατά μήκο ε, του ποταμού. Κυρίως ε, οι τομείς ε, της οικονομικής και εκπαιδευτικής συνεργασίας είναι για μένα σημεία κλειδιά όσον αφορά και την συνεργασία στα, στο μίσο που ανέφερα, θα υποφεληθούν οι άνθρωποι κατά μήκο του ποταμού. Επίσης θα μπορούσε εδώ πέρα να συνεισφέρει, όπως είπα, και η σταδιακή ε, εξομοίωση των πτυχίων με το σύστημα Bachelor και Master, αλλά και διάφορα άλλα αποδειγματά. Επίσης θα ήθελα να εδραιωθεί αυτή η στρατηγική σε όλα τα περιφερειακά μέσα της πολιτικής. Νομίζω πως πρόκειται για το μέλλον ενός τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Για ένα λεπτό. Ο κύριος Ερτουγκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συναδελφοί, αναγκαιότητα ευρωπαϊκών λύσεων και σχεδίων ανάγκης. Νομίζω πως καθίσταται πιο φανερή στους ευρωπαϊκούς ποταμούς που συνδέουν τις ευρωπαϊκές χώρες. Ένα αρνητικό παράδειγμα είναι η στρατηγική, η καταστροφή που έγινε πριν από δύο χρόνια σε μια εξορρυκτική βιομηχανία που βεβαίω εξαπλώθηκε σε ολόκληρο τον ε, Δούναβη και βέβαια οι μεταφορέ εδώ πέρα έχουν ιδιαίτερη σημασία και εγώ ω συγγετής στα διευρωπαϊκά δίκτυα θεωρώ πω η εσωτερική ναυσιπλοεία είναι πάρα πολύ σημαντικό τρόπο μεταφορά γιατί βεβαίω έχει ακόμα πάρα πολύ μεγάλο δυναμικό και είναι φιλική προ το περιβάλλον και βεβαίω αυτό δεν σημαίνει πω πρέπει να γίνει με κάθε τίμημα. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν την προστασία του περιβάλλοντος και αναφέρθηκε πως ένα από τα τελευταία κομμάτια του Δούναβη που ρέει ελεύθερο στην ε, Βαβαρία θα αλλάξει, θα αλλάξει η κήτη του. Αυτό είναι αρνητικό παράδειγμα. Ο υπουργό Δε Περιβάλλοντος της Βαβαρίας το αναγνώρισε αυτό. Θα πρέπει όμως να πείσει και τον Πρωθυπουργό του και τον Ομοσπονδιακό Υπουργό Συγκοινωνιών πως κάθε δεν χρειάζεται άλλη επένδυση σε μελέτες υπενθυμίζω αυτά τα 16,5 εκατομμύρια ευρώ τα οποία έδωσε επιπροσθέτωση η Κομισιόν σε αυτή τη μελέτη τα οποία δυστυχώς είναι πεταμένα λεφτά και θα πήγαιναν καλύτερα σε αυτό το οποίο είπε ο κ. Στόιρερ δηλαδή σε ανταλλαγές των νέων στο Δούναβι. Σας ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Η κυρία Λόχ Μπίλερ ε, έχει μία μπλε κάρτα. Θέλετε να απαντήσετε, κύριε Λόχμπιλερ, έχετε 30 δευτερόλεπτα. Κύριε Ερτούγ, είπατε πως είναι αναγκαίο να έχουμε καλύτερες συγκοινωνίες στην εσωτερική ναυσιπλοεία και αναφερθήκατε και στην προστασία του περιβάλλοντος. Πώς θα λύνατε ε, το ζήτημα αυτό ακριβώς της ε, αλλαγής του, της κήτης του ποταμού. Σας ευχαριστώ κυρία Λοχμπίλερ για το ερώτημα. Πράγματι, στη στρατηγική αυτή υπάρχει κάποια αντίφαση. Αφενός μιλάμε για προστασία του περιβάλλοντος και αφετέρου ε, υποστηρίζουμε τους στόχους αυτών που θέλουν να καταστρέψουν τον Δούναβη. Είναι σαφές, το είπα, δεν επιτρέπεται με κάθε τίμημα να προσπαθούμε να επιτύχουμε την κινητικότητα. Τα πλοία πρέπει να προσαρμοστούν στο ποτάμι και όχι αντιστρόφως. Νομίζω πως μπορούμε να επιτύχουμε τους ε, στόχους που έχουμε, αλλά όπως είπα και η οικολογία είναι εξίσου σημαντική με την οικονομία. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε για την απάντηση και στη μπλε κάρτα. Τώρα μπαίνουμε στη διαδικασία Catch the Eye. και ο κύριος Βιντάλ Κουάδρας ε, θα προεδρεύσει. Ο κύριος Βιντάλ Κουάδρας είναι πολύ πιο άνετος ως προς το χρόνο μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας Catch Γι' αυτό και θα αναλάβει την Προεδρία. Πολλοί ζήτησαν το λόγο και ίσως αυτό οφείλεται στο μέγεθος του Δούναβη. Και γι' αυτό και ενδιαφέρονται τόσο πολύ. Είναι τόσο μεγάλο το ενδιαφέρον. Περνάμε λοιπόν στη διαδικασία Catch the Eye. Ο κύριος Μέσαρος έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Τα τελευταία χρόνια ο Δούναβης έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές και η περιφέρεια αντιμετωπίζει δυσκολίες. Έχουμε καλύτερη συνδεσιμότητα μεταξύ των χωρών της περιφέρειας και της περιφέρειας ε, του Ευξήνου Πόντου η περιφέρεια Ευρώπης και Δούναβη μπορεί να μας βοηθήσει να πετύχουμε οικονομικούς στόχους, καλύτερη ανταγωνιστικότητα, διαχείριση του περιβάλλοντος, αλλά πολλά ακόμα πρέπει να γίνουν. Πρέπει να εξυγχρονίσουμε τα σημεία επαφής του Δουνέβη και να έχουμε καλύτερη πρόσβαση στα μέσα που είναι διαθέσιμα για μας. Καλύτερη λοιπόν πρόσβαση, εναλλακτικέ χρηματοδοτικές πηγές και η ενέργεια πρέπει να διατίθεται με μεγαλύτερη ασφάλεια και σε χαμηλότερη τιμή. Για όλα αυτά χρειάζεται καλύτερη συνεργασία. Ο Δούναβης καλύπτει μεγάλο μέρο Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο συνολικά στη ζωή της Ένωσης γιατί έχουμε δυναμικό και καινοτομία και ε, ε, ανάπτυξης και επιχειρηματικό. Μπορεί να είναι μια σημαντική ε, περιοχή για την Ένωση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σόγκορ έχει το λόγο για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, ο Δούναβης ξεκινάει από το Αδρυμό, Δρυμός και φτάνει στη Μαύρη Θάλασσα περνά από πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων που εντάχθηκαν αργότερα και τις βοηθίζει, βοηθά να φτάσουν το οικονομικό επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι άλλες που θέλουν να γίνουν μέλη. Είναι λοιπόν ένα σύμβολο που ενώνει το δυτικό και το ανατολικό μέρος της Υπήρου. Όσον αφορά τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Δούναβι πρέπει να ενταχθεί στην πολιτική συνοχή. Είναι η υλοποίηση ενός ε, σχεδίου που καλύπτει σημαντικές περιοχές χρειαζόμαστε περιεχόμενο, χρειαζόμαστε συγκεκριμένα έργα στη στρατηγική αυτή που θα είναι επωφελή για τις χώρες, για την κεντρική Ευρώπη, ώστε η κεντρική Ευρώπη να ανακάμψει με καλύτερο τρόπο. Θα πρέπει λοιπόν να αναθεωρήσουμε κάποιες προτεραιότητές μας. Θα ήταν καλό αυτό για να φροντίσουμε να επιτευχθούν αποτελέσματα που μπορούν να βελτιώσουν το επίπεδο ζωής των ανθρώπων που ζουν εκεί. Γι' αυτό ε, εύχομαι κάθε επιτυχία σε όλα τα κράτη-μέλη που αφορά το έργο αυτό. Πιστεύω θα υπάρξει πεδίο συνεργασίας. Ευχαριστούμε κύριε Σόγκορ. Η κυρία Τσικάου έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Με το ψήφισμα της 15ης Φεβρουαρίου 2011 το Κοινοβούλιο ζήτησε από την Κομισιόν να γίνονται περιοδικές διαβουλεύσεις για τον εξυγχρονισμό της στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή του Δούναβη. Η Επιτροπή μας είπε ότι θα δημοσιεύσει την πρώτη έκθεση στην αρχή του επόμενου έτους και ελπίζουμε να επικαιροποιείται κάθε δύο χρόνια. Το Φόρουμ για το Δούναβι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ορίζει από το 2009 σημεία προτεραιότητας και τομείς προτεραιότητες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες δεν έχουν στείλει όλα τα κράτη-μέλη σχέδια για τις καταπροτεραιότητα δράσεις. Έτσι ώστε να υπάρξει επαρκής χρηματοδότηση. Τώρα συζητάμε για το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο μέσα στα πλαίσια του μηχανισμού Connecting Europe. Γι' αυτό θέλουμε να προωθήσουμε και τομεακά σχέδια για την περίοδο 14-20 ως προς τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα θέλαμε μία ξεχωριστή γραμμή για το Δούναβι. Ευχαριστούμε την κυρία Τσικάου. Ο κύριος Πίρκελ. Κύριε Πρόεδρε, Θεωρώ πως πρέπει να δούμε τον Δούναβη πρώτα απ' όλα σε έναν οικονομικό άξονα και με αυτόν τον τρόπο να τον αναπτύξουμε. Γιατί οι επενδύσεις είναι λογικές και αηφόρες όταν υπάρχει μια, μια γενικότερη λογική. Βεβαίως ξεκινάμε τον τομέα της ενέργειας, των μεταφορών μέχρι και του τουρισμού, αλλά όλα αυτά είναι επιτυχημένα μόνο εάν τα έργα αυτά συμβιβάζονται μεταξύ τους. Προτείνω λοιπόν όπως ε, και ε, στα διευρωπαϊκά δίκτυα να οριστεί ένας συντονιστής ο οποίος πραγματικά θα υποβάλει χρονοδιαγράμματα και σχέδια επενδύσεων για να έχουμε πραγματικά στόχους για αυτόν τον δια, τον βασικό διάδρομο στην Ευρώπη και θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Επίτροπο σε ποιο βαθμό βλέπει εδώ πέρα την υλοποίηση του διαδρόμου του Δούναβη που είναι ένας βασικός διάδρομος ε, και την σύνδεσή του με τη στρατηγική για τον Δούναβη. Σας ευχαριστώ. Κύριος Κορτές. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να συγχαρώ την Επιτροπή Ανάπτυξης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την όθηση που έδωσαν στην στρατηγική αυτή. Νομίζω ότι οι στόχοι είναι κατά προτεραιότητα στόχοι όχι μόνο για τους πολίτες ε, της Λεκάνης του Δούναβη, αλλά για όλους τους πολίτες της Ευρώπης. Θα πρέπει να προωθούμε παρόμοιες ε, στρατηγικές όπως στην περίπτωση της Κανταβρίας, δηλαδή να προωθήσουμε παρόμοια σχέδια στον Ατλαντικό. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε αυτές τις μικροπεριφέρειες υπάρχει πολύ ψηλή ανεργία. Ευχαριστούμε κύριε Κορτές. Λουαν. Ο κύριος Λούαν. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, η στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη που προώθησε η Αυστρία και η Ρουμανία οδηγεί σε ευρεία προβλήματα για να είναι καρποφόρα αυτή η στρατηγική και για να υπάρχει η εδαφική, οικονομική και κοινωνική συνοχή σε αυτή την περιοχή θα πρέπει να έχουμε ουσιώδη χρηματοδότηση Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χρηματοδοτικοί πόροι είναι περιορισμένοι και ότι η απορρόφηση είναι ιδιαίτερα περιορισμένη, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες για να βελτιώσουν την απορρόφηση των πόρων και για να προσελκύσουν κεφάλαια από τον ιδιωτικό τομέα. Πρόκειται για ένα ζωτικό τομέα της οικονομίας μας και θα συνεισφέρει στην ευημερία αυτών των λαών για την ανάπτυξη γενικότερα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Πάσκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Η περιφέρεια του Δούναβη προσφέρει μεγάλες ευκαιρίες συνεργασίας για τις χώρες που το περιβάλλουν. Είναι ένα σημαντικός ε, υδάτινος δρόμος που, μεταφέρει, που μεταφέρονται αγαθά από τη Γερμανία στον Εύξηνο Πόντο. Η, οι δάτινες μεταφορές είναι σημαντικές για την προστασία του περιβάλλοντος θεωρούμε ότι θα επέλθουν, ε, θα γίνουν τεχνολογικές αλλαγές ώστε να μπορέσουν να μεταφέρονται περισσότερα αγαθά μέσω του Δούναβη. Πρέπει να δώσουμε σημασία στο περιβάλλον. Οι μελέτες ε, περιβαλλοντικών επιπτώσεων πρέπει να είναι στοιχείο κάθε στρατηγικής που αφορά το Δούναβη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Πάσκα. Ο κύριος Πάνκι έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Ως ούγγρος βουλευτής ε, πρέπει να πω πως ε, είναι θετικό το ότι βρίσκεται αυτό το θέμα στη μερίσια διάταξη του Κοινοβουλίου οι προλαλήσαντες ε, μίλησαν όλοι για τη στήριξή του και θα συμφωνήσω και εγώ. Πρέπει να επιτύχουμε επιτέλους να έχουμε αυτά αποτελέσματα. Ε, αν έχουμε καλύτερες διασυνδέσεις θα έχουμε πάρα πολύ θετικά αποτελέσματα στον τομέα της ανταγωνιστικότητα της δημιουργίας θέσεων εργασία ε, που θα είναι διαρκής. Ο Δούναβης μπορεί να μα βοηθήσει να αναπτυχθούμε όλοι μαζί και δεν υπαρχουν επίση επίσης πάρα πολλά ε, κράτη-μέλη αλλά και χώρε που είναι εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και μπορούμε έτσι να έρθουμε σε επαφή, να συνεργαστούμε, να δουλέψουμε μαζί και αυτό είναι σημαντικό για το μέλλον και την συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και μη κρατών μελών. Επίση, είμαι υπερήφανο ω Ούγγρο για το ότι η κυβέρνησή μα στην Ουγγαρία έχει καταβάλει κάθε προσπάθεια για να στηρίξει αυτό το πρόγραμμα. Και μάλιστα πριν από λίγε εβδομάδε έστειλε ε, μια, ένα κατάλογο στα κράτη-μέλη για μέτρα τα οποία μπορούν να αναλυθούν από εκείνο. Σας ευχαριστώ. Ε, Κάλεμπα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, σήμερα νομίζω πως μπορούμε μετά από ένα χρόνο να αξιολογήσουμε θετικά την στρατηγική αυτή έχουμε 15 εκατομμύρια Ευρωπαίους που επηρεάζονται και έχουμε πάρα πολλά έργα τα οποία έχουν ξεκινήσει ε, και βεβαίως ε, βλέπουμε και στο επίπεδο της διοίκησης ε, των κρατών μελών έχει ληφθεί το μήνυμα αλλά στους ανθρώπους δεν έχει φτάσει ακόμα στην ε, κάτω Αυστρία το Πανεπιστήμιο του Δούναβη είχε κάνει ένα σχετικό συνέδριο και νομίζω πως αυτό είναι αυτό το οποίο πρέπει να γίνει σήμερα, δηλαδή να αναπτύξουμε αυτή τη στρατηγική του Δούναβη, να το αναλάβει και η κοινωνία των πολιτών γιατί θα πρέπει να αναπτυχθεί αυτή η περιοχή όλοι μαζί και επίσης είναι σημαντικό να δούμε πως χρησιμοποιούμε μόνο ένα μικρό κομμάτι του ποταμού, γύρω στο 10% για μεταφορέ. αλλά αυτό επιτρέπει να το κάνουμε μόνο αν σεβόμαστε και την φύση. Σας ευχαριστώ. Και... Η κυρία Μπασέσκου έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η στρατηγική υπέρ του Δούναβη έχει μεγάλη ε, σημασία για μένα διότι από εκεί προέρχομαι, από μία παραδουνάβια περιοχή. Έχει μεγάλη σημασία η οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Θα πρέπει να προωθηθούν υποδομές που θα βοηθήσουν ολόκληρη την περιοχή. Μία από αυτές είναι η γέφυρα που συνδέει την πόλη Καλαφάτ με την πόλη Βιντίν που έχει χρηματοδοτηθεί και θα χρηματοδοτηθεί και το 2013 επίσης η περιοχή του Αγίου Γεωργίου θα προωθήσει τον τουρισμό στο Δέλτα του Δουνάβεως. Θα πρέπει να προωθήσουμε λοιπόν την συνεργασία στην περιοχή. Και ως προς τις χρηματοδοτήσεις πιστεύω ότι ο μελλοντικός προϋπολογισμός θα πρέπει να έχει μία ξεχωριστή γραμμή υπέρ του Δούναβη. Ευχαριστούμε κυρία Μπασέσκου. Τελείωσαμε, τελειώσαμε με τη διαδικασία Catch the Όλοι έλαβαν το λόγο και προέρχονταν Ε, από χώρες της Αυστρο-Ουγγρικής Αυτοκρατορίας που διετέλεσαν ε, υπό τους Αψβούργους. Τώρα έχετε εσείς το λόγο, κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Απελευθερώθηκα από τα ακουστικά μου. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση αυτή. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στα τέσσερα βασικά θέματα που έθεσαν. Την διαχείριση και τη χρηματοδότηση, μεταφορές και περιβάλλον, διαφάνεια, δημοκρατικός έλεγχος και ε, αντιμετώπιση των νέων και φυσικά η διαδικασία υλοποίηση και υποβολή εκθέσεων. Θέλω όμως καταρχήν να ευχαριστήσω όλους σας για τις παρεμβάσεις σας, γιατί σπάνια βρίσκει κανείς τόσο ε, ευρία υποστήριξη για ένα κοινό έργο. Πιστεύω ότι όλοι σας πιστεύετε ότι η Ευρώπη χρειάζεται τη στρατηγική του Δούναβη και ότι η στρατηγική του Δούναβη έχει πολλά ακόμα να προσφέρει. Μόλις αρχίζουμε να συνειδητοποιούμε τις δυνατότητες του τι μπορεί να επιτευχθεί μέσω αυτών των, ε, της, αυτής της περιφερειακής προσέγγισης όπως είπε και ο πρόεδρος. Είναι η κοινή ιστορία μας, το κοινό μας παρελθόν αλλά και το κοινό μας μέλλον θεωρώ εγώ. Επιτρέψτε μου να συνεχίσω με τα ερωτήματα του κυρίου ε, Μάτουλα Ματώη και Τόπουλα όσον αφορά το περιβάλλον. Αυτό που έχει σημασία είναι να επιτευχθεί καλή λύση στις διαπραγματεύσεις 22 και 3 Νοεμβρίου και αργότερα για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο με το Κοινοβούλιο. Αυτό θα είναι μόνο η αρχή. Αν θέλουμε να πετύχει αυτή η προσπάθεια θα είναι πολύ σημαντικό να είναι πολύ στενή η συνεργασία με τα κράτη-μέλη, με τις περιφέρειες και να δουλέψουμε για το σχεδιασμό. Να σχεδιάσουμε μαζί ποια θα είναι τα βασικά έργα που θα γίνουν υπό την αιγίδα της στρατηγικής του Δούναβη. Αυτό που θα βοηθούσε πολύ θα ήταν να υπάρξουν κεφάλαια ήδη από τώρα διαθέσιμα για τα έργα. Έτσι ώστε να πούμε αυτό είναι ο κατάλογο των έργων προτεραιότητα. αυτά είναι σημαντικά για την περιφέρεια, αυτά θα θέλουμε να υλοποιηθούν και να χρηματοδοτηθούν μέσω των, ε, του Διαρθρωτικού και Ταμείου και του Ταμείου συνοχή στο επόμενο διάστημα. Αυτό το οποίο θα προσπαθούσαμε να κάνουμε στην Επιτροπή είναι να χρησιμοποιήσουμε το ότι ήδη από τώρα η προσέγγιση αυτή έχει συμπεριληφθεί στο σχέδιο κανονισμού για τι πολιτικέ συνοχή. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να ενταχθούν σε ένα κοινό στρατηγικό πλαίσιο στις συμβάσεις εταιρικής σχέσης και στο συντονισμό. Ο κύριος Στόρεν Ματούλα ρώτησε πώς θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εμπλακεί περισσότερο στην προετοιμασία και το σχεδιασμό. Θεωρούμε ότι αυτό μπορεί να γίνει με την συμμετοχή μας στη σύνταξη της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και την διαχείριση του κοινού πλαισίου. Όπως προέκυψε και από τη συζήτηση, θεωρώ ότι σε πολλά κράτη-μέλη οι δυνατότητες απορρόφησης της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης δεν είναι και οι καλύτεροι και θεωρώ ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά με την καλύτερη διαχείριση αυτών των πόρων, με συνέργειες και την προσφορά επιπλέον τεχνικής βοήθειας προς τα κράτη-μέλη που σαφώς έχουν προβλήματα απορρόφησης των διαρθρωτικών ταμείων. Θεωρώ ότι σε αυτό πρέπει να επικεντρωθούμε και μέσω των νέων χρηματοοικονομικών κανονισμών που προδίνουν νέε δυνατότητες απλούστευση όλων αυτών των διαδικασιών. Μπορούμε σαφώς να πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον. Τώρα όσον αφορά το περιβάλλον και τις μεταφορές. Αυτό είναι πάντοτε ένα σοβαρό ζήτημα. Εξισορρόπηση των περιβαλλοντικών ε, ζητημάτων με τις ε, ανάγκες της περιοχής. Ένα ε, σημαντικό υδάτινο δρόμο όπως είναι ο Δούναβης. Πρέπει να υπάρξει ε, ανεξάρτητη ε, συμμετοχή εμπειρογνωμόνων. Πρέπει όμως και η Επιτροπή να προσπαθήσει να συμβιβάσει τα περιβαλλοντικά ζητήματα με τις ανάγκες της, ε, δια, ε, της πλεύσης στον Δούναβη. Θα πρέπει λοιπόν τα περιφερειακά κοινοβούλια και οι πολίτες να εμπλακούν στις συζητήσεις αυτές. Όχι μόνο από αυτή τη σκοπιά, αλλά και από τη σκοπιά του τι μπορεί να πετύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω μιας καλής ε, εφαρμογής της στρατηγικής του Δούναβη σε συγκεκριμένες περιοχές. Επίσης αναφέρθηκε ότι πρέπει να στραφούν περισσότερο προς τους νέους. Πράγματι γιατί υπάρχει υπάρχει ανεργία ε, ε, σε ολόκληρη την Ευρώπη και οι νέοι μπορούν να υποφεληθούν από αυτά τα προγράμματα. Θεωρώ ότι οι τομέα προτεραιότητας υπαριθμών 7 ακριβώς σε αυτό επικεντρώνεται. Πώς μπορούμε δηλαδή να φέρουμε τα πανεπιστήμια ε, σε συνεργασία μεταξύ τους, να θεσπίσουν κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα και προγράμματα διδακτορικών διατριβών ε, για τους νέους. Όλα αυτά πιστεύω θα αποτελέσουν πολύ καλή ευκαιρία ώστε οι νέοι να γνωριστούν καλύτερα αλλά και να ε, επιδιώξουν και να βρουν περαιτέρω ευκαιρίες σπουδών και εργασίας. Όσον αφορά τώρα το ζήτημα που ετέθη για τον Δούναβη και τις προτεραιότητες των αξώνων. Πράγματι είναι στο δίκτυο τέν ο Δούναβης και θα θεωρηθεί ως άξονας προτεραιότητας, έργο προτεραιότητας στο επόμενο ε, πολιετές δημοσιονομικό, ε, στην επόμενη δημοσιονομική προοπτική. Επίσης ε, ε, μας ερώτησαν πώς θα σας ενημερώνουμε για το τι έχει γίνει με αυτή τη στρατηγική. Όπως σας είπα, αυτή τη στιγμή κάνουμε την αξιολόγηση της πρώτης χρονιάς. Πώς εφαρμόστηκαν τα πράγματα το τελευταίο αυτό διάστημα και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η έκθεση θα είναι έτοιμη πολύ πριν από τον επόμενο Ιούνιο. Ε, θα χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία μας για την επόμενη περίοδο και θα δούμε εκ των υστέρων τι θα μπορούσε να είχε γίνει καλύτερα κατά την τρέχουσα περίοδο. Άρα μπορούμε να εμπνευστούμε για τα νέα έργα, τις νέες δραστηριότητες που θα ξεκινήσουμε στις τα πλαίσια της στρατηγικής του Δούναβη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Περνάμε στο επόμενο θέμα που είναι η έκθεση που αφορά το διαμεσολαβητή. Κυρία Ματσόνη, έχει το λόγο για τέσσερα